Χαίρετε κυρία Γεωργίδα. Euh, euh, Ευχαριστώ. Άρχεται η συζήτηση λοιπόν. Το λόγο έχει επίτροπος η κυρία Κρέτσου. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ιδιαίτερη χαρά σας απευθύνω το λόγο εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή τη φορά. Ανταποκρίνομαι στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για δήλωση σχετικά με την ευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία κατά κύριο λόγο φορά δύο κυβερνήσεις, του Ηνωμένου Βασιλείου και της ε, Ιρλανδικής Δημοκρατίας, που εδώ και σειρά ετών έχουν στενά συνεργαστεί για ε, την ειρήνη από τον Δεκέμβριο του 1993. Ε, αμέσως καλωσόρισε τη δήλωση η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεσμεύτηκε να προχωρήσει για κοινωνική και οικονομική πρόοδο στην περιφέρεια και με χρηματοδότηση προγραμμάτων από τη Διορθωτικά Ταμεία. Έκτοτε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα και τα συμβουλευτικά ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ειρηνευτική διαδικασία. Για μένα αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό γιατί η ίδια η Ένωση είναι επιτυχημένο παράδειγμα ε, επιτυχούς συμφιλίωσης. Το 1994, αμέσως μετά την διακήρυξη ε, των παραστρατιωτικών ε, οργανώσεων στη Βόρεια Ιρλανδία ότι επέρχεται πλήρης κατάπαυση του πυρός και βίας, ο Ζακ Τελόρ, τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διατράνωσε την πλήρη προσήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ευτική διαδικασία με ισχυρή υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείναμε ένα νέο πακέτο για να προχωρήσει η συμφιλίωση και η κοινωνική και οικονομική ανοικοδόμηση. Αυτό ε, ήταν μια καινοτόμο δράση και πρόγραμμα ειρηνευτικό, το οποίο εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη το 1995 και κάλυπτε τη Βόρειο Ιρλανδία και ε, τις ε, ε, παραμεθόριες κομιτείες της Ιρλανδίας που κατοικούν 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι. Μέχρι το 2013 ήταν 1,3 δις ευρώ σε τρεις γύρους η χρηματοδότηση και 2 δις από τα κράτη-μέλη. Ε, χρησιμοποιήθηκαν με διαφορετικό τρόπο, με κοινοτικά επιτόπου προγράμματα ε, στο κοινωνικό τομέα για κοινή ε, συνεργασία για να ξεπεραστεί η κληρονομιά του παρελθόντος. Ήταν μακροπρόθεσμη αυτή η περίοδος, τώρα Έχουμε μια νέα που αρχίζει 2014-2020. Κοινοβούλιο και κράτη-μέλη συμφώνησαν για ένα νέο ειρηνευτικό πρόγραμμα. 230 εκατομμύρια ευρώ θα είναι τα κοινοτικά χρήματα, συν 40 περίπου από τα κράτη-μέλη. Αξιότιμα μέλη, αυτά τα προγράμματα έχουν πετύχει σε μεγάλο βαθμό και είναι πολύ σημαντικό στοιχείο στην ευρύτερη νευτική διαδικασία που σας είπα αφορά δύο κράτη-μέλη κατά κύριο λόγο και κατά πρώτο λόγο. Πάντα αναγνωρίζαμε ότι το πρόγραμμα αυτό δεν ε, ε, ε, χωράει εύκολες λύσεις. Είναι στρατηγικό, έχει βάθος χρόνου και μακροπρόθεσμη συνεργασία, εταιρική σχέση για να οικοδομηθεί η συμβίωση και η διασυνοριακή συνεργασία. πολύ θετική ήταν η επίδραση στην ε, πράξη επιτόπου και στη Βόρεια Ιρλανδία και στις παραμεθόριες ε, κομιτείες ε, της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι συνεργάζονται για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και έχουν μπει τα θεμέλια για ένα κοινό μέλλον. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα έργα αυτά βοήθησαν να αλλάξει η στάση και η συμπεριφορά του κόσμου. Σκέφτονται τα ίδια τους ε, τα προβλήματα της προκαταλήψης, αρχίζουν να ανέχονται το διπλανό τους και να χτίζουν μια νέα κοινωνία. Το πρόγραμμα, ας πούμε, ε, έχει εστιάσει στη δημιουργία θετικών σχέσεων σε τροπικό επίπεδο. Να καταλάβει ο κόσμος τι έχει γίνει στο παρελθόν, να το επεξεργαστεί και να το ξεπεράσει. Πάνω από 5.000 ε, άνθρωποι έχουν συμμετάσχει σε εργαστήρια για το ξεπέρασμα της σύγκρισης, πάνω από, της κρίσης, συγγνώμη, πάνω από 7.000 ε, ε, δέχτηκαν βοήθεια για μετατραυματικό σοκ και ψυχολογική υποστήριξη. Αυτά προετοιμάζουν το έδαφος για την επόμενη γενιά έτσι ώστε οι νέοι να έχουν και τις ικανότητες και τις δεξιότητες που χρειάζονται αλλά και την στάση για να αποφεύγεται η διαθρησκευτική βία. Θα πρέπει ε, η νευτική διαδικασία να γίνει κτήμα του λαού εκεί. Θα πρέπει να ερθαρρυνθεί ο κόσμος να βρει τις ίδιες λύσεις του για τα προβλήματα. Ξέρουμε ότι ε, πρόσφατα υπήρξε κάποιο πιστοδρόμηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε την απόφαση να συνεχίσει τη χρηματοδότηση στην περίοδο 14 με 20 και αναγνώρισε ότι υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει και δεν έχει τελειώσει η υπόθεση. Όπως γνωρίζουμε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014 και με 2020 ε, καθυστέρησε όπως και το ρυθμιστικό συνολικό, το κανονιστικό Υποβλήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου ε, το πρόγραμμα από τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει τις παρατηρήσεις της. Στο νέο πρόγραμμα θα δημιουργηθούν ευκαιρίες για τους νέους της Βορείου Ιρλανδίας και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τους νέους πρέπει να βοηθήσουμε για να δούμε μια κοινωνία πιο ανεκτική αύριο που να μπορεί να εγκαταλείψει το μίσος και τη βία του παρελθόντος και εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και ακόμα και τα ευαίσθητα και τα καθόδη ζητήματα θα αντιμετωπίσουμε και θα παραμείνουμε ε, στο πλευρό του νέου προγράμματος παραστάτες. Είναι σημαντικό να θυμίσουμε ότι το ειρηνευτικό πρόγραμμα δεν είναι μόνο οικονομικής φύσεως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει γενικότερα την ειρηνευτική διαδικασία με 350 εκατομμύρια 20 ε, χρόνια ε, στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία και τη συμφιλίωση. Και από το 2007 επίσης, από τότε που άρχισαν να λειτουργούν οι θεσμοί και ο κύριος Μπαρόσο ε, έκανε μια ε, υπηρεσιακή ομάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μελετά όλες τις δυνατότητες από κάθε σκοπιά κάθε πολιτικής. Η Task Force λοιπόν για τη Βόρεια Ιρλανδία εργάζεται υπό τη δική μου ευθύνη πλέον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περιφερειακή πολιτική ε, έχει διευρυνθεί και σήμερα απαρτίζεται από εκπροσώπους 18 γενικών διευθύνσεων της Κομισιόν και παίζει ρόλο στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη με την ευρύτερη έννοια. Πολλοί από εσά θα είδατε την έκθεση που εκδώσαμε αρχές του μηνός ε, και περιγράφουμε τις ε, δραστηριότητες της Task Force την επταετία που λειτουργεί. Είναι, ήταν θετική η αντίδραση και χαίρομαι γι' αυτό. Αναγνωρίστηκε και ο ρόλος ε, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Ιρλανδίας Ρόμπερτσον και, Ρόμπινσον συγγνώμη, και από τον ε, Αντιπρόεδρο τον Μάρτιν Μαγκίνες. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένω να ακούσω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Οι πολιτικές ομάδες. Πρώτος ο κύριος Κέλλη από το ΕΛΚ. Δύο λεπτά. Ως εισηγητής στο ίδιο θέμα την προηγούμενο χρόνο και επικεφαλής της αντιπροσωπείας μου στο ΕΛΚ έχω την τιμή να παρουσιάζω αυτό το ψήφισμα για την ειρηνευτική διαδικασία και θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω την πρώην συνάδελφό μας την κυρία Επίτροπο. Χωρίς αμφιβολία η ειρηνευτική διαδικασία στην Ιρλανδία θα μπορούσε να θεωρηθεί θαύμα διότι οι άνθρωποι που μισούσαν ο ένας τον άλλον και που έβγαζαν εύκολα πιστόλι, τώρα κάθονται στο τραπέζι λόγω της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής. Και γι' αυτό πρέπει να ευχαριστήσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κύριος Νίκολσον που ήταν εδώ όλα αυτά τα χρόνια μπορεί να το πιστοποιήσει. Υπάρχει όμως και ένα αδιέξοδο, το λέω αδιέξοδο και όχι τέρμα της διαδικασίας, ελπίζουμε ότι αυτό το ψήφισμα θα ενθαρρύνει όλες τις πλευρές να συνεννοηθούν με ανοιχτό πνεύμα και εδώ δεχτήκαμε πριν από μερικές εβδομάδες τον ε, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και μετά τον κύριο Νέσμοντ όλοι μας είπαν και οι δύο μας είπαν ότι πρέπει η Ευρώπη να σώσει τη Βόρεια Ιρλανδία. Αυτό είναι το πνεύμα του ψηφίσματος γιατί ο λαός της Ιρλανδίας θέλει την ειρήνη. Είδα και εγώ με τα μάτια μου τι γίνεται, τι προσπάθειες γίνονται και τι προβλέπεται για τα επόμενα ένα-δύο χρόνια. Θέλει ο κόσμος να συνεχίσουν οι προσπάθειες, άρα πρέπει όλες οι πολιτικές πλευρές να συνεννοηθούν με βάση αυτό το ψήφισμα για να υποστηρίξουμε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κέλλη. Υπάρχει γαλάζια κάρτα, τη δέχεστε, κύριε Κέλλη μου. Δέχεστε γαλάζια κάρτα. Κύριο Σέφριτς. Και εμείς κύριε Κέλλη στην ομάδα μου θέλουμε να προχωρήσουν τα πράγματα Υπάρχουν όμως και δύο προβλήματα του παρελθόντος και ελπίζω να συμφωνήσουν όλοι. Το Μπέρμιχαμ είναι στην εκλογική μου περιφέρεια και οι οικογένειες της υπόθεσης των 21 δεν έχουν ακόμη δικαιωθεί. Εσείς συμφωνείτε να κλείσει και αυτή η υπόθεση και να δικαιωθούν αυτές οι οικογένειες. Ναι, υπάρχουν θέματα κληρονομιάς από το παρελθόν Μερικά από αυτά έχουν λυθεί τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίσουν να επιλύονται. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι τμήμα της όλης ειρηνευτικής διαδικασίας. Για να βλέπει ο κόσμος και τι έγινε, αλλά και πώς μπορεί η ειρήνευση να οδηγήσει σε διόρθωση των πραγμάτων. Δεν αρκεί απλώς να κρίνουμε εδώ στο Κοινοβούλιο, να καταδικάζουμε και να επιβραβεύουμε, αλλά εφού όλοι θέλουν ειρήνη, θέλουν όλοι και δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ και τώρα για τους σοσιαλδημοκράτες ο κύριος Μωράης δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς όρισε είναι Επίτροπος η οποία ήταν στις τάξεις της πολιτικής μας ομάδας ε, και έχουμε επίσης ε, το κοινό ψήφισμα που πρόθεσε η πολιτική μας ομάδα και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό μια που όλοι εδώ θέλουμε να υπάρχει μια οφαστικότητα όσον αφορά τη, αυτό το, το πρόβλημα της Βορειοϊρλανδίας και να εφαρμοστεί η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Αυτό το κοινοψήφισμα μας υπενθυμίζει αυτά τα οποία διαπιστώσαμε. Πρόκειται για ένα παράδειγμα προς μίμηση για επίλυση κρίσης. Ε, είναι μια ειδική περίπτωση, είναι κάτι ιστορική σημασία για το Ηνωμένο Βασίλειο, και την ε, Ιρλανδία. Πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή. Αυτό αφορά και τον κύριο Νίκολσον, γιατί συνεργαστήκαμε με τα Ιρλανδικά και Βορειοϊρλανδικά κόμματα, με το Sinn Féin, με ε, θέμα την συμφιλίωση και έχουμε επομένως ε, ως στόχο την συμφιλίωση. Αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε και αυτό κάνει και το ψήφισμα είναι να επιλύσουμε τα επιμέρους προβλήματα, να σημειωθεί πρόοδος για το βαροελλανδικό ζήτημα. Δεν θα πρέπει να ε, το ξεχάσουμε ή να το ε, υποτιμούμε. Έχουμε τις διαπραγματεύσεις που είναι δύσκολες, μεγάλη διαδικασία και θα πρέπει επομένω να σημειωθεί πρόοδος, να έχουμε ένα παράδειγμα προς μίμηση επίλυση διαφορών. Αυτή η διαδικασία ε, ειρήνευσης θα πρέπει να διέπεται από αλληλοκατανόηση να ξέρει ο καθένας, ο άλλος τι προσδοκά και τι θέλει, τι ελπίζει και έτσι θα πρέπει ομένω να τεθεί ένα τέρμα σε αυτή τη σύγκρουση και θα πρέπει ο καθένας να καταλάβει και να μπει στη θέση του άλλου. Συμβιβασμός χρειάζεται. Αυτό είναι ε, η πολιτική τέχνη του συμβασμού και είναι πολύ σημαντικό ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως μας εξήγησε η Επίτροπος. Είμαστε περήφανοι για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συνεχίσουμε να βοηθούμε για την επίλυση του προβλήματο. Πρόεδρο, Σα ευχαριστούμε αγαπητέ συνάδελφε. Και τώρα τον λόγο έχει ο κύριο Νίκολσον για 1,5 λεπτό για το ECR. Σα ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, επίσης επιτρέψτε μου να πω καλώς όρισε η Επίτροπο στο Κοινοβούλιο ε, περιμένουμε πώς και πώς να συνεργαστούμε μαζί σας και ελπίζουμε πραγματικά τώρα που αναλάβατε το χαρτοφυλακείο σας να έρθετε και να ξανέρθετε και να δείτε ε, επιτόπου στην Ιρλανδία τι πρόοδος έχει σημειωθεί. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβεβαιώσει το ότι συνεχίζει να υποστηρίζει την Ιρλανδία. Ε, τη Βόρεια Ιρλανδία είναι επίσης του προβλήματος, γιατί έγινε τόσες δεκαετίες. Είχαμε μια μειονότητα η οποία ε, σημείωσε αυτό το πρόβλημα, αλλά ο λαός εκεί αυτό το οποίο θέλει είναι να χτίσουμε μια καλύτερη κοινωνία. Βλέπουμε ότι με τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθά στην αυτή διαδικασία και έχουμε όλες αυτές τις ε, γενιές ε, προγραμμάτων ειρήνευσης, έχουμε την και έχουμε όλα τα σημάδια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να πετύχει βήματα πρόοδου στην Βόρεια Ιρλανδία. Α καταλάβουμε ότι αυτή η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε την Task Force η οποία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Ακριβώς ε, όπως υποσχέθηκε και δεσμεύτηκε η Επίτροπος κυρία Κρέτου. Να μην ξεχνούμε ότι σε κάποια φάση πριν από κάποια χρόνια ο κόσμος θεώρησε ότι έχει κλείσει το, το θέμα. Αυτό δεν είναι αλήθεια, οπότε θέλουμε και χρειαζόμαστε την βοήθειά σας. Και τώρα, λέει τον λόγο έχει η κυρία Χάρκιν για 1,5 λεπτό για τους φιλελευθέρους. Χάρκιν. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να ευχηθώ καλώς όρισε η νέα Επίτροπος ξανά στο Κοινοβούλιο. Ποιος είναι ο βασικός ε, στόχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλαμε να φτιάξουμε την οκτώτα για να σταματήσουν οι πόλεμοι, για να βρεθούν κάποιοι ε, τρόποι, μέθοδοι συνδύωσης. Και για πάρα πολλούς, ιδίω για εκείνους που δεν θυμούνται τον πόλεμο, ίσως αυτό φαίνεται κάτι απλό, απλοϊκό, σαν ε, στόχος. Και αυτό γιατί γεννήθηκαν και ζουν μέσα στην ειρήνη κάθε μέρα. Ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί. Αλλά όμως δεν είναι κάτι αυτονόητο το ότι υπάρχει ειρήνη. Ποτέ δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι κάτι το οποίο ολοκληρώθηκε, πετεύθηκε για πάντα. Είναι μια διαδικασία. Και αυτό ισχύει ε, μια ολόκληρη διαδρομή και για την Ευρώπη και για την Βόρεια Ορλανδία. Οπότε ε, αυτή η διαδρομή βρίσκεται μόνο στην αρχή της στην Βόρεια Ορλανδία. Χρειάζεται επομένω αρρωγή αυτή η προσπάθεια μπορεί ανα πάσα στιγμή να καταρρεύσει ή να ανατραπεί. Οπότε ε, θα πρέπει όποτε έχουμε κάποιο πίσω γύρισμα να την στηρίζουμε, να την ξαναστείλουμε στα πόδια και να συνεχίζουμε. Έχει βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει χρηματοδοτήσει ένα σωρό προγράμματα, τα δύο τελευταία δε είχαν ως προτεραιότητα τη συμφιλίωση των κοινοτήτων και ε, της κοινωνίας γενικότερα και έχουμε τα νέα ταμεία ή τους νέους πόρους που θα καλύψουν τους νέους και τους ανηλίκους. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο για το πώς θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ε, παιδείας και εκπαίδευσης. Θα είναι αυτό μια καλή αρχή. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει για 1,5 λεπτό εξ ονόματος της ΚΟΕ Κύριε κυρία Άντερσον. Ο Μάρτιν Μακίνες πριν από λίγο καιρό μας ενημέρωσε ε, και την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο ο πρόεδρος Σούλτς έκανε μια δήλωση για την ετοιμότητα και την προθυμία του Κοινοβουλίου μας να βοηθήσει. Όπως λέει και το ψήφισμα, η εφαρμογή της συνευτικής διαδικασίας έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Καλούνται όλα τα μέλη να εργαστούν επικοδομητικά προς μια βιώσιμη λύση της σύγκρουσης και πλήρη υλοποίηση της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής και της επόμενης συμφωνίας. Καλωσορίζω τη χτενισινή επίσκεψη ε, των ε, εκπροσώπων ε, ε, των ενωτικών. Ε, η ειρνευτική διαδικασία έχει υποστηριχθεί και από τη Task Force του Μπαρόσο, πρέπει να συνεχιστεί και η χρηματοδότηση και ο Ντελόρ, Βουλφ Μάτις, Χούμπνερ, Χάν και τώρα εσείς κυρία Κρέτσο όλοι αυτοί οι επίτροποι συνεισφέρουν και σας βοηθώ. Είναι σημαντική συνεργασία μεταξύ ευρωβουλευτών από έξι πολιτικά κόμματα. Ε, με ευθύνη δεσμευόμαστε να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Το ψήφισμα θα πρέπει να αντανακλά ε, και τα όσα πιστεύουν οι κυβερνήσεις και ε, τα ενεχόμενα μέρη. Συνέχεια της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής. Ξέρω ότι η συμφιλίωση θα χρειαστεί καιρό, αλλά πιστεύω ότι κάποτε θα έρθει όταν όλοι ε, θα συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο μαζί θα κερδίσουμε, αλλιώς θα χάσουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τέλερ έχει το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Τέλερ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ε, πολλοί εκτός της Ιρλανδίας θεωρούν ότι έχουν τελειώσει οι συγκρούσεις και οι ταραχές όταν παραδόθηκαν τα όπλα και κηρύχθηκε η κατάπαυση του πυρός, δεν σημαίνει ότι έχει έρθει ειρήνη. Είναι πολύ δρόμος και μακρύς. Η ειρνευτική διαδικασία πάντα θα χρειάζεται αναζωογόνηση και συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση. Ε, ε, στο Belfast μόλις μετακόμισε ε, η οικογένεια του γαμπρού μου και είδα ποιες είναι οι εγκληματικές δραστηριότητες και η βία που υποβόσκει. Και αυτά φαίνεται περνάνε παρατήρητα ή αναπάντητα. Αυτές οι αντικοινωνικές ε, δράσεις ε, είναι και εγκληματικές και οφείλονται στην ανεργία και στην οικονομική δυσπραγία και όχι σε οικονομικές, ε, πολιτισμικές ή θρησκευτικές διαφορές θα πρέπει να κερδίσουμε τα μυαλά και τις καρδιές των ανθρώπων, να τους ε, αποσπάσουμε από τη βία. Υποστηρίζω πραγματικά αυτό το ψήφισμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Νάταλ. Για ένα λεπτό. Κυρία Επίτροπε, ο δυτικός κόσμος προχτές μόλις ε, ε, γιόρτασε την πτώση του τείχους του Περολίνου. Στο Μπέλφαστ έχουμε ακόμα τείχη που χωρίζουν τις δύο κοινότητες. Ε, ποια είναι η ευημερία. Μπορεί να μην υπάρχει βία. 1,7 ε, δις στερλίνες λογαριασμό έχει να πληρώσει το Ηνωμένο Βασίλειο και ενώ έδινε 100 εκατομμύρια ε, το Υπουργείο Οικονομικό μας στη Βόρεια Ιρλανδία για να βγάλει το χρόνο. Είναι η μεγαλύτερη ενεργεία από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, λοιπόν, αντί να δίνουμε κάθε μέρα 55 εκατομμύρια στερλίνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προτείνω αυτά τα λεφτά να τα δίνουμε στη Βόρεια Ιρλανδία που τα έχουν πικρά ανάγκη. Συμφωνούμε όλοι γι' αυτό και καλό είναι. Αλλά έχουμε αφήσει την ε, Βόρεια Ολλανδία ε, στη μοίρα της, σε μια οικονομική έρημο μετά από αυτό το βίο πόλεμο. Ε, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδική Δημοκρατία, Αμερικανή, Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχαν οικονομικά να εξασφαλίσουν βιώσιμη ειρήνη. Απομένουν ακόμα πάρα πολλά να γίνουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Ντότσο. Α, υπάρχει γαλάζια κάρτα. Προς τον κύριο Νάταλ, τη δέχεστε, δέχεστε τη γαλάζια κάρτα. Ε, Ο κύριο Μπροκ. Μα κύριε Λούταλ, Νούταλ δεν τρέπεστε καθόλου. Η εσωτερική σας πολιτική δίνεται λάθος οικονομικά στοιχεία. Χρησιμοποιείτε για εσωτερική προπαγάνδα υποχρεώσεις σας, για τη χώρα σας, ε, για την ενευτική υποτίθεται διαδικασία όπου έπαιξε πολύ καλό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και εδώ να χρησιμοποιείτε την ευτική διαδικασία για να κάνετε εσωτερική προεκλογική εξατία στη χώρα σας, είναι, τι να πω, δεν ε, εξυπηρετεί το σημαντικό ε, αυτό της ειρήνης. Είναι πολύ φτηνά αυτά τα λόγια και τα επιχειρήματα. Χωρίς μικρόφωνο, κύριος Νάταλ. Μα κοιτάξτε, είναι απλά τα πράγματα. Είπε η Επίτροπος, 350 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτό είναι 6 μέρες από συνεισφορά που δίνουμε εμείς στο Ευρωπαϊκό ε, ε, ε, Κουρβανά από το Ηνωμένο Βασίλειο. Να φύγετε, λέει ο Μπρόκ, με χαρά να φύγω. Γιατί η χώρα μου θα είναι πιο ελεύθερη, πιο δημοκρατική και πιο ευήμερη. Από εδώ που είναι εγκλωβισμένη σε αυτή τη διεφθαρμένη οργάνωση το βασικό είναι η νευτική διαδικασία η οποία προχωρεί. Αλλά οικονομικά η Βόρεια Ιρλανδία είναι σε τέλμα. Και αν εξοικονομήσουμε χρήματα που δεν θα δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούμε να επενδύουμε στη Βόρεια Ιρλανδία ακόμα περισσότερα. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ε, και τώρα το λόγο έχει. Σύμφωνα με τον κατάλογο, η κυρία Ντότς. Για 1,5 λεπτό, παρακαλώ. Yes. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, κυρία Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση επί πολύ καιρό ήταν, από πολύ καιρό είναι φίλος της Ιρλανδίας και χαίρομαι γιατί mm. σήμερα λέει ότι θα συνεχίσει την υποστήριξή της και τους επόμενους μήνες. Η Βόρεια Ιρλανδία εκτιμά ιδιαίτερα αυτή τη βοήθεια την εποχή που αρχίζουμε να χτίζουμε μια πιο ευημερούσα και πιο ειρηνική κοινωνία. Τα πρόσφατα χρόνια θελήσαμε να περάσουμε όντως σε μια πιο ειρηνευμένη κοινωνία. Οι τρομοκράτες απέτυχαν και όλοι και οι ενωτικοί βασίζονται σε αποκλειστικά ειρηνικούς στόχους πλέον στο Κοινοβούλιο. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι η πολιτική θα κερδίσει με στόχο μόνο τη δημοκρατία για να υπάρξει μια πιο ευημερούσα και ειρηνική Βόρεια Ιρλανδία με σταθερότητα. Η λειτουργία των δημοκρατικών μας θεσμών είναι κάτι βασικό για την οικοδόμηση αυτής της νέας πραγματικότητας. Όλες οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις λένε ότι υπάρχει μεγαλύτερη υποστήριξη για να μείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο η Βόρεια Ιρλανδία περισσότερο από ποτέ στην ιστορία μας. Και μάλιστα αυτή η υποστήριξη βασίζεται <clears throat> στην ύπαρξη των δύο παραδόσεων. Ε, υπάρχει και στις δύο παραδόσεις στη Βόρεια Ιρλανδία. Και η λειτουργία της ίδιας της δημοκρατίας τα προβλέπει όλα αυτά από την πλευρά των ενωτικών τουλάχιστον θετικά θέλουμε να απλοποιηθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων και να υπάρξει καλή διαχείριση και, διαχείριση και διακυβέρνηση στη Βόρεια Ιρλανδία. Υπάρχει γαλάζια κάρτα, την δέχεστε, από τον κύριο Τάνοκ. 30 δευτερόλεπτα κύριε μου. Χωρίς, χωρίς μικρόφωνο. Mm. Ναι, δουλεύει, δουλεύει, εντάξει. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Ντότζ, είπατε ότι τώρα υπάρχει πολύ μεγάλη υποστήριξη για την παραμονή της Βόρειας Ιρλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά αν ο κύριος Νάτολ κάνει αυτά που θέλει, τότε θα φύγει η Βόρεια Ιρλανδία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα συμφωνούσε αυτό με την πολιτική των καθολικών στο Δουβλίνο και πώς θα άλλαζε αυτό την πολιτική σας. Με μικρόφωνο παρακαλώ. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Είπα ότι υπάρχει μεγαλύτερη υποστήριξη για να παραμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο η Βόρεια Ιρλανδία γιατί το βασίζω σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει ανεξάρτητα στη Βόρεια Ιρλανδία και δείχνει ότι περισσότεροι Ιρλανδοί ταυτίζονται με το Ηνωμένο Βασίλειο και περισσότεροι θεωρούν τον εαυτό τους Βόρειο Ιρλανδό. Είναι ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει καμία επιθυμία για την επανένωση της Ιρλανδίας. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει, τουλάχιστον σε λίγο χρόνια, και ότι μόνον αν γίνει κάτι τέτοιο θα γίνει μόνο με βάση τη δημοκρατική θέληση του λαού, πράγμα το οποίο δεν το βλέπω. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκονζάλης Πόνς, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαιρόμαστε για την κατάσταση αυτού του ψηφίσματο που έχει στόχο να προωθήσει μια διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία που φαινόταν να είχε αποτολματωθεί. Ω κοινωνία οφείλουμε να προωθούμε την ειρήνη, αλλά και ω κοινωνία επίση έχουμε και την ηθική υποχρέωση να μην λησμονούμε τι συνέβη και όταν συνέβη ήταν τρομακτικό. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τι έγινε στη Βόρεια Ιρλανδία και για ποιο λόγο ήταν οι δολοφονίες, γιατί οι δολοφονίες ήταν ε, ε, εξ ονόματος θρησκειών στις οποίες εμείς πιστεύουμε οι Ευρωπαίοι και για ευρωπαϊκές αξίες. Η σύγκρουση ήταν ένοπλη, σύραξη που άφησε πολύ βαθιές ουλές και τραύματα που ακόμα δεν έχουν κλείσει και θα αργήσουν να κλείσουν. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την ευτική διαδικασία και να απομονώσουμε τους ακραίους και να προωθήσουμε την κατανόηση. Αλλά δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι αν δεν έχουμε υπόψη μας τι έγινε, τα θύματα ε, θα πληρώσουν τελικά τα σπασμένα, όπως πάντα πληρώνουν τα θύματα την τρομοκρατία. Το είπε η Επίτροπος και έχει δίκιο ότι αυτό αφορά αποκλειστικά και μόνο τη Βόρεια Ιρλανδία. Αλλά θα θέλαμε να έλεγε εμείς οι Ισπανοί ε, στο κείμενο να μην νοείται ε, ατιμορρησία. Όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη πληρώνουν δύο φορές τα θύματα. Στη Βόρεια Ιρλανδία ήταν χιλιάδες τα θύματα από την ένοπλη σύραξη. Αλλού, χωρίς ένοπλη σύγκρουση, ε, αλλά με ειρήνη, υπάρχουν επίσης χιλιάδες θύματα της τρομοκρατίας. Χρειάζεται ένας ευρωπαϊκός χάρτης των δικαιωμάτων των θυμάτων και να ζητήσουν συγνώμη οι τρομοκράτες να πληρώσουν, να εκτίσουν την ποινή τους και να βοηθήσουν οι τρομοκράτες ε, στη διαλεύκανση όλων των εγκλημάτων. Και όλοι οι υπόλοιποι με τιμή και αξιοπρέπεια να ποτίσουμε ένα φόρο τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, η ατιμορρησία είναι ένας δεύτερος θάνατος για τα θύματα, εάν γλιτώνουν οι τρομοκράτες. Δεν νοείται ατιμορρησία στον κόσμο που να μπορεί να ευσταθεί, ούτε στη Βόρεια Ελλανδία. Σε αυτό το ψήφισμα, κυρία Πρόεδρε, δεν υπάρχει καμία αναφορά στα θύματα της τρομοκρατίας. Απίστευτο είναι και προλαβαίνουμε ακόμα να το διορθώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Ραμόν το για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, στα ισπανικά μιλώντας, θα, μόνο αυτό θα έπρεπε να αποτελεί σεβασμό στο τι γίνεται στην Ιρλανδία. Γιατί έμεσα αυτό σημαίνει υπενθύμηση και σεβασμό αυτού που έλεγε η Ιντήρα Γκάντι, ότι δηλαδή δεν υπάρχει ένας δεδομένος δρόμος για την ειρήνη. Ο τρόπος είναι η ειρήνη. Είναι μια διαδικασία, διαδικασία δύσκολη όπως και την Ιρλανδία και θα πρέπει να βοηθήσουμε πρόβλημα για όλη την Ευρώπη. Να βοηθήσουμε και άπαξ και όλοι οι Ιρλανδοί εδώ συμφωνούν. Αυτό είναι φανταστικό, είναι υπέροχο. Θα πρέπει επομένως να προσέξουμε ότι αυτή η δύσκολη και μακρά διαδρομή προς την ειρήνη ε, επιδέχεται βοήθεια, επιδέχεται το να λέμε την αλήθεια, απαιτεί το να κάνουμε μια συμφιλίωση, να μην περιθωριοποιούμε κανέναν και θα πρέπει και η Βόρεια να έχει ε, οικονομική ενίσχυση. Ε, ότι δηλαδή περνάει αυτή τη δύσκολη διαδρομή και ότι οι συμβίωση που επιδιώκουμε εκεί επιδέχεται τη βοήθεια της Ευρώπης. Αυτό έχει γίνει ε, σαν προσπάθεια και στην χώρα των Βάσκων. Είναι σημαντικό να βοηθήσει η Ευρώπη και οπότε και εμείς θα πρέπει να αναζητήσουμε και πάλι συνένεση των ε, Ιρλανδών βουλευτών εδώ όλων, ούτω ώστε να συνεχιστεί αυτή η δύσκολη πορεία για την ειρήνευση. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να υποστηρίξω εγώ που δεν είμαι Ιρλανδός, αλλά που μου αρέσει να πηγαίνω στην Ιρλανδία. Χτες ε, το βράδυ θυμηθήκαμε την κατάπαυση του πυρός στο Dixmount, ε, που ξέρετε είναι στη Φλάνδρα, in Flanders Fields, που είναι το σύμβολο του ματέου του πολέμου και είναι και σύμβολο της ε, συμφιλίωσης, της ειρήνης, του διαλόγου, της ειρηνικής επίλυσης. Και αυτό μας οδήγησε τελικά και στην ειρήνευση στην Ιρλανδία. Και με μεγάλο θαυμασμό κοιτάξαμε από τη Φλάνδρα ε, το θάρρος και των Ιρλανδών και των Βρετανών για να καταλήξουν στη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα ε, χειροκροτούσε, αλλά δυστυχώς ποτέ δεν είναι αυτονόητη η ειρήνη. Και τώρα τα εμπόδια που ορθώνονται και είναι και απειλές αρχίζουν να μας ανησυχούν θα πρέπει να συνεχίσουμε να προωθούμε τη βιώσιμη ειρήνη. Στην Ευρώπη όλοι ενδιαφερόμαστε να επιτύχει αυτή η διαδικασία στην Ιρλανδία και θα πρέπει να είναι υπόδειγμα για άλλες συγκρούσει ε, που δεν έχουν επιληθεί και εκτός της Ευρώπης και εντός και εδώ σκέφτομαι τη χώρα των Βάσκων προκειμένου που δεν έχει επιληθεί ακόμα αυτή η υπόθεση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κάθριν Μπέρντερ έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ορίζετε κυρία Επίτροπε. Ο λαός της Βορειοϊρλανδίας έχει περάσει πάρα πολλά από τότε που είναι η συμφωνία του το 97 γιατί τις Μεγάλες Παρασκευής άφησαν πίσω τους τη Δία και τώρα υπάρχουν πολιτικά θεσμικά όργανα, υπάρχουν εκπρόσωποι όλων των ε, κομμάτων και το είπε ο, ο, ο ο καλύτερα έτσι πάρα πολύ. Και οπότε τώρα στην Ιρλανδία προχωρούμε προς την ειρήνευση με μεγάλα βήματα από τα άτομα, από τους φορείς, από αυτή την διερημένη συμφωνία, ώστε να υπάρχει μια ε, αντεκτική, βιώσιμη ειρήνη. Ακόμη υπάρχουν βέβαια προβλήματα, ούτω να μην μπορούμε την ενευκή Συμφωνία να την εφαρμόσουμε 100%. Θα πρέπει αυτά τα προβλήματα να επιληθούν. Συνεχίζει το διχασμό της κοινότητε παρά τι ε, προσπάθειε που γίνονται προ το αντίθετο, ιδίω όσον αφορά στέγαση, όσον αφορά τα σχολεία. Ε, οι νέοι οφούνται στο έγκλημα, αντικοινωνική συμπεριφορά, γίνονται και πολλές πράξεις βανδαλισμού. Όμως θα πρέπει να τους βοηθήσουμε αυτούς τους νέους ανθρώπους και αυτό το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχει ρόλο πάρα πολύ σημαντικό για την συμφιλίωση μεταξύ των κοινοτήτων. Και την επόμενη πενταετία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει ούτως ώστε να τεθούν οι βάσεις για μια βιώσιμη ειρήνη. Επίση, η οικονομική ανάπτυξη βοηθά την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει όλου του εμπλεκόμενου να του ευχαριστήσουμε για αυτά τα προγράμματα, για αυτέ τι προσπάθειε. Ε, να συμφιλειωθούν οι κοινότητε, να δοθούν ε, ελπίδε, ευκαιρίε, προγραμματισμό, συνεργασία και έτσι να βοηθήσουμε ούτω ώστε να υπάρχει μια ε, αδιαίρετη κοινωνία για όλου στη Βορειοελλανδία. Σα ευχαριστούμε πολύ. Νίριάντα τώρα. Δεν ξέρω κάτι υπάρχει ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο. Κύριε Πρόεδρε, η διαδικασία της ειρήνευσης αναγνωρίζεται παντού ως ε, έμπνευση, ως ελπίδα. Ιδίω για εκείνους που προσπαθούν να επιλύσουν άλλες, τις δικές τους σύγκρουσεις. Άρα θα πρέπει αυτή τη διαδικασία να την υποστηρίξουμε και να επιλύσουμε τα προβλήματα που ακόμα υπάρχουν όλες οι συμφωνίες. Θα πρέπει επομένως ε, να εφαρμοστεί ο νόμος για την ε, Ιρλανδική γλώσσα τα κελτικά και επομένως ε, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την άγνοια, την μη κατανόηση για την κουλτούρα, τον πολιτισμό, την ισότητα και δυστυχώς οι προτάσεις χάς δεν έγιναν αποδεκτές. Πραγματικά καλή προσπάθεια ήταν αυτή, αλλά μπορεί να βοηθήσει το Κοινοβούλιο. Να βοηθήσουμε τη διαδικασία και να αποκτήσουν όλοι στην Βόρεια Ιρλανδία μέλλον. Τώρα η κυρία Εύανς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε. Το 12 η Ευρωπαϊκή Ένωση κέρδισε το βραβείο Νόμπελ και διαβάζω γιατί για εδώ και 60 χρόνια προώθησε την ειρήνευση και τη συμφιλίωση, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη. Πολλοί τότε είχαν σαρκάσει, αλλά πιστεύω ότι η Διεθνώς Ένωση έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο ειρηνευτικό. Παρά πολλά καλά βήματα που έγιναν τελευταία, όμως η ειρηνευτική διαδικασία στην Ιρλανδία έχει ακόμα δρόμο να διανύσει. Έχουν κατορθωθεί πολλά για την περάτωση της βίας και για τη συνεννόηση των μερών αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ακόμη έχει επιτευχθεί μια βιώσιμη ειρήνη. Χρειάζεται πολύς χρόνος και πολλή προσπάθεια. Και γι' αυτό το λόγο τα ειρηνευτικά προγράμματα της Ένωσης και το ειδικό task force της Κομισιόν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει λοιπόν και το Κοινοβούλιο να δείξει ότι έχει τη θέληση να στηρίξει την ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κλούν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και κυρία Επίτροπη για τη δήλωσή σας που τόνισε τη χρηματική στήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Βόρεια Ιρλανδία. Είχα την ευχαρίστηση να επισκεφθώ την Ιρλανδία για να δω με τα μάτια μου την αξία αυτών των χρηματοδοτήσεων για κοινοτικά, δικοινοτικά προγράμματα, ιδίως για τη στήριξη νέων που υπήρξαν θύματα της βίας για οποιονδήποτε λόγο, από οποιαδήποτε μεριά ψυχολογικής ή σωματικής βίας. Πολλούς που φυλακίστηκαν, καταδικάστηκαν. Υπάρχουν λοιπόν πολλά θετικά που έγιναν στην Ιρλανδία και είναι ευχάριστο να το βλέπει κανείς. Αυτή την εβδομάδα στο Belfast εντατικοποιούνται οι συζητήσεις και είναι και αυτό θετικό. Υπάρχουν ακόμη αδιέξοδα, αλλά δεν αφαιρεί αυτό τίποτα από την αξία των προσπαθειών που έχει γίνει, που γίνει με την κυβέρνηση, από την κυβέρνηση της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και που θα ωφελήσουν όλο το λαό της Ιρλανδίας. Η συνέχιση των προσπαθειών θα χρειαστεί φυσικά να μιλήσει και για το παρελθόν και την κληρονομιά που μας άφησε. Θέλω να αναγνωριστεί η προσπάθεια που έγινε και να καταλάβουν όλοι ότι έχουμε πάρα πολλά να κερδίσουμε αν συνεχίσουμε να συνεννοούμαστε και πάρα πολλά να χάσουμε αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Θα συνεχίσουμε ελπίζω να προχωράμε και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την υποστήριξή τους Ζητώ δε από όλους τους συμπαλόμενους να κάνουν, να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ντάνς για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ποτέ δεν θα φανταζόμουν να μου πει κάποιος δική μου είναι η χώρα, όχι η δικιά σας. Τι είναι αυτά που λέτε κύριε Νάταλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες γιατί ανακατεύονται και χειραγωγούν τις καταστάσεις ε, οι βουλευτές ε, των εργατικών συμφωνούν ε, να εφαρμοστεί το συντομότερο στο σύνολό της η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Με τεράστια χαρά και προνόμιο εργάστηκα για τον Υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Ιρλανδίας όταν στην στηνόντουσαν οι θεσμοί και τα όργανα και η δικαιοσύνη. Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια. Άξιζε τον κόπο όμως. Και ένα βασικό στοιχείο αυτής της επιτυχίας ήταν να καταλάβουμε ε, ότι διακυβεύονται ζητήματα για όλους, για τον τρόπο με τον οποίο ε, χειριζόμαστε τις τύχες μας. Μια νέα γενιά έχει μεγαλώσει και δεν θα πρέπει να γνωρίσει κανένα ε, μίσος και να μην φοβάται ούτε τις βόμβες ούτε τις σφαίρες κανείς. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Η διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία μπορεί να δείξει στον κόσμο τα ωφέλη της πολιτικής για την ειρήνη. Ακούστηκε το, το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει. Δεν θα πρέπει να συνεχιστεί, γιατί θα αποθαρρυθούν οι νέοι ηγέτες. Θα πρέπει η νέα γενιά να καταλάβει ότι είναι απείρως προτιμότερη η πολιτική από την άλλη εναλλακτική λύση. Θα πρέπει να έρθεις να καθίσεις σε ένα τραπέζι και να συζητήσεις με τον πολιτικό σου αντίπαλο και πολιτικά και συναισθηματικά και οικονομικά να συμμετέχουν οι πάντες και είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι της Ευρώπης ε, η Ιρλανδία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δέχεστε μια μπλε κάρτα. Έχει ερώτηση συνάδελφος. Παρακαλώ. Θα ήθελα επ' ευκαιρία ο κύριος Νίκολσον να ευχαριστήσω ε, τον κύριο Ντάνς. Ήταν πολύ χρήσιμη. Δέχεται από πλευράς μου να του πω ότι ο λαός της Βόρειας Ιρλανδίας είναι βαθύτατα ευγνώμονες για τη βοήθεια που τους δίνει το Κοινοβούλιο. Ποτέ ε, δεν ε, ε, έδρασαν μονομερός και μεροληπτικά. Και κύριε Μπρόκ έχετε δίκιο, γιατί έφυγε ο κύριος Νάταλ τώρα, αλλά εγώ δεν είμαι καθόλου πεπισμένος ότι τα λεφτά αυτά θα τα στέλνει η Βρετανική κυβέρνηση στη Βόρεια Ιρλανδία. Για να δούμε τι θα γίνει. Να διορθώσω και κάποια άλλα πράγματα. Θέλω εδώ να αποτίσω φόρο τιμή στο Ζακ Ντελόρ απόψε και στην δόκτωρα Μόνικα Βούλφ Μάτις που ήταν η πρώτη επίτροπος για περιφερειακές υποθέσεις και προώθησε αυτή την ευτική διαδικασία και είναι ένα ουσιαστικότατο κομμάτι όλης αυτής της ειρηνευτικής προσπάθειας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρος. Και τώρα θα παρακαλούσα όλους τους βουλευτές όταν ζητούν να κάνουν ερώτηση με την μπλε κάρτα να κάνουν ερώτηση για να μπορέσει ο ερωτώμενο να απαντήσει. Τώρα κύριε Ντάν, θέλετε να απαντήσετε, δεν έγινε ερώτηση, ήταν τοποθέτηση αυτή. Ναι, όντως δεν έχω να απαντήσω τίποτα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής. Ομιλήτρια, κυρία Ζητγάνσκα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, παρά την υπογραφή της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής. Τώρα ε, βλέπουμε διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις και βιοπραγίες. Γι' αυτό θα πρέπει να επανακινήσει η ενευτική διαδικασία, να λυθεί το συντομότερο αυτή η σύγκρουση. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να ε, πατάξουμε τη βία. Υποστηρίζω πλήρως το ψήφισμα και είμαι πεπισμένη ότι η ειρευτική διαδικασία θα μπορέσει να προχωρήσει. Τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν όχι μόνο την οικονομία και την κοινωνία να αναπτυχθεί στη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά θα εξασφαλίσουν και ένα ασφαλές και ε, ε, μερών μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Πίτσουλα. Ένα λεπτό. Uz dobrodošlicu povjerenici želio bih u raspravi Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω ότι γίνονται πολλές ε, συμφωνίες σημαντικές και η συμφωνία του Ντέιτον και του Ερντούτ που θυμάστε ε, ήταν ε, το τέλος του πολέμου στη Βοσνία Ζεγοβίνη από τη χώρα που προέρχομαι κι εγώ. και η συμφωνία του Ερντούτ έφερε και την ένταξη ορισμένων εδαφικών Χωρί χωρίς όμως η συμφωνία του Ντέιτον να δημιουργήσει ένα κράτος που να λειτουργεί σωστά. Ε, στην Κροατία ε, η περιοχή γύρω από το Δούναβι έχει ε, υποστεί μεγάλες ζημίες και τελικά για την αποκατάσταση της ειρήνης και μετά την αποκατάσταση της ειρήνης έχει ε, επιστρέψει ο σερβικός πληθυσμός. Ε, θεωρώ μια αντίστοιχη κατάσταση έχουμε στη Βόρεια Ιρλανδία. Η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής είναι πάρα πολύ χρήσιμη και θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ταραμπέλα έχει το λόγο. Πρόεδρε, κυρία Επίτροπη, θέλησα να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση γιατί σήμερα όταν ακούμε ότι υπάρχουν θρησκευτικέ κοινότητε ή άλλε κοινότητε που δεν ανέχονται μία την άλλη, αυτό είναι, συμβαίνει στη Βαγδάτη. Όταν ήμουν 10 χρονών και έψαχνα την επικαιρότητα, ακούγαμε συχνά London Derry και Belfast από πόλεις. Ε, χαίρομαι που δεν μιλάμε πάρα πολύ για αυτές τις πόλεις πια, γιατί η νευτική διαδικασία ε, στέφθηκε με επιτυχία μέχρι σήμερα. Υπόθηκε προηγουμένως μία μειονότητα θέλει να ξαναρχίσουν οι σειράξεις. Γι' αυτό εμείς οφείλουμε βεβαίως να υποστηρίξουμε το ψήφισμα αλλά και τη διαδικασία που είναι και μακρά και δύσκολη. Και θα ήθελα τελειώνοντας να πω ότι η ειρήνη δεν είναι ποτέ δεδομένη ε, θα πρέπει πάντα να αρχίζουμε από την αρχή, να υφαίνουμε στον αργαλιό ξανά και ξανά. Στη Βόρεια Ιρλανδία υπάρχει ένας κατευνασμός ε, και αντιδράσαμε γιατί ήταν απαράδεκτο, γιατί είναι δίπλα μας, βέβαια είναι διπλανή χώρα, αλλά είναι δική μας. Και γι' αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θαυμάσια και ελπίζω να πάνε στη σωστή κατεύθυνση και να μην ξαναρχίσουν οι σειράξει παρά ε, κάποια πολεμοχαρή που ακούμε από μεμονωμένους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται η συζήτηση αυτή ε, με βάση τον κατάλογο των ομιλητών και περνούμε στη διαδικασία Catch the Eye, αυθόρμητες τροποθετήσεις. Η κυρία Μαγκίνες έχει το λόγο. you, Ευχαριστώ κύριε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε γιατί τονίσατε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ηρευτική διαδικασία στην Ιρλανδία. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που δεν είναι από την Ιρλανδία και που έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι υπάρχει λέξη αδιέξοδο στο ψήφισμα, αλλά δεν υπάρχει λέξη τερματισμός των συνομιλιών. Είναι απλώς ένα αδιέξοδο. Και υπάρχει πολιτική ευθύνη των συμβαλωμένων των δύο μερών στην Ιρλανδία και στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας και το Ηνωμένο Βασίλειο για να βγούμε από το αδιέξοδο. Εγώ μεγάλωσα κοντά στα σύνορα με την μεξή Βορείο Ιρλανδίας και Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και καθημερινά άκουγα τρομερά πράγματα για δολοφονίες παιδιών, μητέρων, πατέρων. Τα παιδιά μου όμως δεν γνωρίζουν αυτή την Ιρλανδία και δεν θέλω ποτέ να επιστρέψει. Είναι λοιπόν σημαντική η συζήτηση και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστούμε. Κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ και εγώ με την υποστήριξη για το ε, ψήφισμα γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη, στην επανόρθωση, στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων, στο διάλογο και στην συμφιλίωση για να μπορούμε να λύνουμε τις βίες συγκρούσεις. Αξιολογώ θετικά την ευρωπαϊκή εμπλοκή σε αυτή τη διαδικασία γιατί συνάδει με τις βασικές αξίες της Ένωσης και αναγνωρίζει ότι μια αιστεία αστάθεια στην Ευρώπη δεν είναι ποτέ αμυγό εσωτερικό ζήτημα, αλλά είναι πάντα ευκαιρία για αλληλεγγύη και συνεργασία μεταξύ όλων, για να βοηθήσουμε να λυθεί το θέμα. Γι' αυτό ο πρόεδρο ε, της χώρας των Βάσκων, η Νίκο Ορκούλιου, συνεργάζεται με ένα πρόγραμμα ε, από την Ιρλανδία για να δανειστούμε από την εμπειρία του και να κλείσει στη χώρα των Βάσκων το θλιβερό κεφάλαιο τη βία. Ζητώ από τα θεσμικά όργανα τη Ένωση να ενδιαφερθούν εξίσου και να εμπλακούν και για στη χώρα των Βάσκων όπως και στην Ιρλανδία και να γίνουν φίλοι του Εουσκάδη της χώρας των Βάσκων γιατί και εμεί το χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ο, ο κύριος ε, Αρίστη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρόταση ψηφίσματος. Ο κύριος Χωρίστη ε, θα πρέπει να εφαρμοστεί στο σύνολό του και ό,τι δεν έχει ε, γίνει ε, να εφαρμοστεί στην Βόρειο-Ανατολική Ιρλανδία. Ευχαριστώ την κυρία Κρέτσου για την προθυμία της και για τη βοήθεια από την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Είπε ότι θα ασχολείται με τα ε, δύσκολα θέματα της συνευτικής διαδικασίας. Η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εκ των όνων κάνευ προς την επίλυση των πολιτικών συγκρούσεων που υπάρχουν ακόμα στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Η πρόταση ψηφίσματος με την οποία συμφωνούν ποικίλε πολιτικές ομάδες μας λέει τα πράγματα με το όνομά τους και καλεί όλα τα μέρη του Κοινοβουλίου να κοιτάνε την κατάσταση και την πραγματικότητα κατάματα για να μπορούμε να τη λύνουμε. Μόνο έτσι. Και δεν μπορώ παρά να ενθαρρύνω και το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εμπλακούν και να συνεισφέρουν με τον ίδιο τρόπο στην ειρήνη και στην ε, επίλυση του προβλήματος στην εουσκαλερία, στη χώρα των Βάσκων. Θα είναι προς όφελος όλων. Ευχαριστώ πολύ. Έθελες. Thank you. λόγο κύριε. Θα ήθελα να εκφράσω το θαυμασμό μου για όλους τους Ιρλανδούς πολιτικούς από κάθε πτέρυγα εδώ που επιδεικνύουν οριμότητα και δύναμη χαρακτήρα ούτως ώστε να μπει στην άκρη ε, αυτή η απέσια σύγκρουση για να πάμε ξανά σε μια καινούργια αρχή. θα πρέπει να αποθεί δικαιοσύνη, θα πρέπει ο κόσμος να μάθει τι γίνεται, αν μη τι άλλο. Και ενώ για την ομάδα των 21, τι έγινε, για αυτούς κατηγορήθηκαν για τις βόμβες στον Πέρμιγκαν, πέρασαν 40 χρόνια. Ακόμα ο κόσμος δεν ξέρει τι έγινε με τους συγγενείς, με τους συγγενείς τους και κανείς δεν βγαίνει να πει την αλήθεια. Σας παρακαλώ, όλους εσάς τους καλούς ανθρώπους της Ιρλανδίας, τους καλούς πολιτικούς, Πέστε μου, πέστε μου τι έγινε με τους 21. Θα πρέπει να κλείσει αυτός ο φάκελος. Πραγματικά εύχομαι καλή επιτυχία. Ο Θεός μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Η κυρία Ντότς. Μα μιλήσατε. Δεν μπορείτε να ξαμιλήσετε τώρα και ε, μπλε κάρτε και τέτοια πράγματα στη διαδικασία κάτι Μιλήσατε προηγουμένω κανονικά στη συζήτηση. Δεν μπορούμε να σας ξαναδώσουμε το λόγο. Λυπούμε και σας ζητώ να με συγχωρήσετε γι' αυτό. Ο κύριος Γιάκοψης, τελευταίος. Μύρε, νέμα αλτερνατίβε, αλτερνατίβε, različitost življenja ευχαριστούμε πολύ. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Μόνη λύση είναι η ειρήνη και ο διάλογος. Υπάρχουν διαφορές. Οι διαφορές όμως είναι δύναμη, είναι πλεονέκτημα, αλλά και η ανεκτικότητα είναι το ίδιο ένα πλεονέκτημα. Ξέρετε ότι εκεί που κατοικούσα είχαμε πόλεμο και δεν υπήρχε ανοιχτικότητα για τα γλωσσικά. Όμως ο κόσμος βρήκε το θάρρος να γεφυρώσει τις διαφορές και έκανε πάρα πολλά η Ευρώπη για την Βορειο Να, ποιος είναι ο αυτού του ψηφίσματος. Θέλουμε να πούμε ένα μπράβο σε αυτούς που βρήκαν το θάρρος να δώσουν, να προσπαθήσουν τόσα πολλά ανοχή, ανεκτικότητα. Έτσι θα πετύχουμε την ειρήνη. Είμαι υπέρ του ψηφίσματος. Η Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφοι, σας ενημερώνω ότι έχουμε μία πρόταση ψηφίσματος. Και πριν αρχίσει η συζήτηση, θα πρέπει να συγχαρούμε και να ευχαριστούμε καλώς όρισε η Επίτροπος για το νέο της καθήκοντα. Ήταν ε, ε, αντιπρόεδρος εδώ, τώρα έχει την Επιτροπή. Έχετε το λόγο κυρία Κρέτου. Πρώτα πρώτα να σας πω πόσο θεωρώ θετικά όλα όσα είπατε και να ευχαριστήσω γενικότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οποία τοποθετούμε στην σημαντική αυτή συζήτηση όπως τονίσατε οι περισσότεροι το ειρηνευτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα πρόγραμμα της Ένωσης ε, στα πλαίσια των διαρθωτικών ε, ταμείων διαρθωτικής ε, πολιτικής και έχετε δίκιο ότι δεν θα πρέπει να στεριώσει η ειρηνευτική πορεία και αυτό προϋποθέτει βέβαια η οικονομική ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης αυτό και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το πρόγραμμα, να έχουμε κάποιες προοπτικές, θετικές, κυρίως για τους νέους, γιατί θα πρέπει να σταθεροποιηθεί η οικονομία και επίσης θα πρέπει να ξανασταθεί στα πόδια της, να ανασυγκροτηθεί και όπως είπατε περισσότεροι είναι πάρα πολύ οδυνηρό να διαπιστώνουμε ότι την 25η επέτειο της πτώσης του τείχου Έχουμε ένα τείχος Βορειοϊρλανδία που στο Μπέλφαστ χωρίζει τις δύο κοινότητες. Βεβαίω και έχουμε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο βοηθάει. Ε, είδαμε πόσα χρόνια, 60 χρόνια πόσο έχει βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να συμφιλιώσει ε, και γι' αυτό και θεωρούμε ότι οι Βορειοϊρλανδοί ηγέτες καθώς και η Ιρλανδική όπως και η Βρετανική κυβέρνηση θα πρέπει να υπολογίζουν ε, στην αμέριστη συμπαράσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη δική μου προσωπικά για να επιληθούν ό,τι προβλήματα ακόμα υπάρχουν και να υπάρχει βιώσιμη ειρήνη. Βεβαίω και πρόκειται να επισκεφθώ τη Βορειοϊρλανδία στο εγγύς μέλλον. Για μένα είναι προτεραιότητα, αλλά και για την Επιτροπή. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το πρόβλημα της χώρας των Βάσκων αυτό το οποίο κάποιοι βουλευτές ετώνησαν και επιτρέψτε μου να σας μιλήσω στην λατινογενή μου ε, μητρική γλώσσα προς τους Ισπανούς συναδέλφους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργεί αιτήσει των κυβερνήσεων. Για την Ιρλανδία υπάρχει αίτημα από Ιρλανδική κυβέρνηση και Βρετανική κυβέρνηση. Όμως, όσον αφορά το βασικό θέμα, δεν έχει γίνει τέτοιο έτοιμο. Εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε να διευκολύνουμε όσον αφορά τις προσπάθειες ειρήνης των δύο πλευρών και σας τονίζω ότι η Επιτροπή πραγματικά θέλει να βοηθήσει, να εξυγχρονίσει την βασική οικονομία με την πολιτική συνοχής να βοηθήσουμε για καινοτομία, ή ε, Το Μπιλμπάο σχεδόν ανασυγκροτήθηκε 100%. Ξαναχτίστηκε με ευρωπαϊκούς πόρους. Πολύ σύγχρονη πόλη σήμερα. Δημιουργήσαμε εκεί βιώσιμες θέσεις απασχόλησης. Task Force για τη χώρα των Βάσκων θέλουμε να γίνει, αλλά θα πρέπει να υπάρχει επίσημο αίτημα προς το Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει σε τελευταίο Μα Μας απευθύνει σύσταση και εμείς συγκροτούμε την Task Force. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζει στα αγγλικά. Πρώτη φορά έρχομαι εδώ υπό αυτή την ε, ιδιότητα και είναι κάπως παράξενο το αίσθημα αυτό να αλλάζω θέση ούτως υπήρ. Πάντως σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε και για το έργο σας και για την τοποθέτησή σας εδώ την Παρθενική υπό τη νέα σας ιδιότητα. Καλή δύναμη και ό,τι επιθυμείτε. Λοιπόν, θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι έχω λάβει ένα κοινό ψήφισμα που υπογράφουν έξι πολιτικές ομάδες και τώρα κλείνω τη συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Και θα περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα, σύμφωνα με την ημέρησια διάταξη. Είναι δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και είπα της εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα